Η κατάσταση λοιπόν είναι ε, σοβαρή, αλλά ε, σας έχω και καλές ειδήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει έξι ψηφίσματα. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση γι' αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την επόμενη συζήτηση. Η οποία αφορά το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα. Και θα δώσω το λόγο στους συντάκτες. Πρώτος ο κύριος Τάνοκ.

Κύριε Πρόεδρε, το σκάνδαλο αναγκαστική άμβλωση ε, στην Κίνα είναι πραγματικά σοκαριστικό. Η Φέγκ Τζιαμέη απήχθη ε, από τοπικού υπαλλήλου ε, στην περιοχή Σενγκζιά και ενώ ήταν 7 μηνών αναγκάστηκε σε άμβλωση. Καταδικάζω τη βαρβαρικότητα αυτή, όπω και όλη η ομάδα μου, και πρόκειται για μια πράξη που ξεσήκωσε κατακραυγή και στην Κίνα, κάτι ασύνηθε. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο τη αναγκαστική άμβλωση λόγω τη πολιτική του ενό παιδιού στην Κίνα παρά ε, τι εκκλήσει για την αποτροπή αυτών των αποτρόπαιων πρακτικών. 118 πρέπει να είναι άρενα και 100 ε, θύλα τα βρέφη τα οποία γεννιούνται και έχει ανατραπεί ισορροπία με τις ε, πρακτικές αυτές. Υπάρχουν αυτές οι πρακτικές οικογενειακού προγραμματισμού. Θα πρέπει όμως προτεραιότητα να είναι η ε, κατάργηση της αναγκαστικής άμβλωσης και αναγκαστικής στήρωσης και στο επόμενο στάδιο του διαλόγου μας με την πρέπει να το θέσουμε κατεπηγόντως στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκο. Κύριος Πέτερλε. Το ψήφισμα človekovo dostojanstvo nedotakljivo. primer splava na kitajskem v katerega je bila prisiljena dvaindvajset letna ženska v sedmem mesecu nosečnosti je dejstvo ki zahteva. Πέτρελε, έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. Ε, περιμένετε μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Να ξαναρχίσω από την αρχή. Περιμένετε, λέει, και μετά ναι, ξαναρχίστε. μου λένε να σας πω να συνεχίσετε να μιλάτε για να ελέγξουμε αν λειτουργούν τα μικρόφωνα καταστάσεις. Λοιπόν, όπως έλεγα, αυτό το ψήφισμα βασίζεται σε μια θεμελιώδη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζεται στο άρθρο 1 για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα αξιοπρέπεια συγκεκριμένα που είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα. Η αναγκαστική άμβλωση μιας 22χρονης γυναίκας στην Κίνα είναι ένα γεγονός το οποίο χρήζει της ε, μέση προσοχής μας. Οι, οι αναγκαστικές αμβλώσεις στην Κίνα πρέπει να καταδικαστούν, διότι είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλούμε την Κίνα να αναθεαρίσει την πολιτική του ενός παιδιού και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι θα πρέπει το θέμα των αναγκαστικών αμπλώσεων να το συμπεριλάβει στις συνομιλίε που έχει με την Κίνα. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν για ποιο λόγο και πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Τα χρήματά τους πρέπει να δαπανούνται μόνο σύμφωνα με τις αξίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε. κύριος Ρωμέβα ή Ρουέντα. Για 1,5 λεπτό. Yes, uh, the facts... Τα... Στις 22 Ιουνίου μια γυναίκα απήχθη, οδηγήθηκε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και της έκαναν ανάβλωση. Ε, η έρευνα η οποία έγινε κατέληξε στο ότι της επιβλήθηκε η άβλωση. Χάρη όμως ε, στην εκστρατεία μέσω του διαδικτύου, αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα έχει περιοριστεί. Αυτή όμω η περίπτωση που ανέφερα προηγούμενα, σύμφωνα με το ε, σχέδιο δράση του Διεθνού Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, όπου αναφέρει ότι υπάρχει δυνατότητα σε κάθε ζεύγο καθώ και σε μονομένα άρμα να καταλήγουν σε ελεύθερε, υπεύθυνε και τεκμηριωμένε αποφάσει για τεκνοποίηση και να διατίθεται πλήρε φάσμα ασφαλών, αποτελεσματικών και υποδεκτών μέθων, μεθόδων οικογενειακού προγραμματισμού και τη επιλογή του. Δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτό καμία μορφή εξαναγκασμού. Καταδικάζουμε λοιπόν την ε, τακτική αυτή και την πρακτική αυτή. Καταδικάζουμε επίση και την απόφαση για την αναγκαστική άβλωση της κυρίας Φέγγ. Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε την συζήτηση που διεξάγεται με ακαδημαϊκούς για την πολιτική περί ενός και μόνο δικού τέκνου. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχάκε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Την περασμένη εβδομάδα από το διαδίκτυο έμαθε ο κόσμος ότι μια γυναίκα έγκυος 7 μηνών, Φένζι Μέι, απήχθη και αναγκάστηκε να κάνει άμβλωση. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός απομονωμένο. Η εμβριοκτονία και η βρεφοκτονία ε, καθώς και οι ε, μαζικές αμβλώσεις για επιλογή του φύλου λαμβάνουν χώρα στην Κίνα ως συνέπεια της πολιτικής του ενός παιδιού. Οι επιλεκτικές αμβλώσεις έχουν αλλάξει και τη δημογραφία. 40 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 40 εκατομμύρια κορίτσια λείπουν. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι ελεύθερος να κάνει την επιλογή του για τον οικογενειακό προγραμματισμό, αν θέλει να κάνει παιδιά, αν δεν θέλει όχι, με τρόπο ασφαλή και οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού είναι λάθος και αυτό κυρίως αφορά γυναίκες έτσι στοχευμένα. Είναι σημαντικό όλες οι γυναίκες να έχουν το θεμελιώδη δικαίωμα της πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία, ε, τη βοήθεια, ε, τη φροντίδα των παιδιών και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Ε, η οργάνωση του ΟΗΕ για τις γυναίκες αρχίζει να ερευνά συστηματικά τι γίνεται στην Κίνα. Και θα ήθελα να πω ότι το γεγονός αυτό που ευτυχώς πυροδότησε μεγάλη συζήτηση και στην Κίνα και στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα του διαδικτύου που επέτρεψε στην ιστορία αυτή να κυκλοφορήσει. Οπότε να τονίσουμε και την ελευθερία του διαδικτύου και να καταπολεμήσουμε τη μαζική λογοκρισία και στην Κίνα. Ευχαριστώ κυρία Σάκε. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βερζιά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το δικαίωμα κάθε γυναίκας ε, για αυτοδιάθεση του σώματός τους είναι θεμελιώδη Το να ε, χρησιμοποιούμε αυτό το δικαίωμα για λόγους ε, πολιτικούς δεν νομίζω ότι σεβόμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά με την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών οι γυναίκες προσπαθούν να αγωνιστούν και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να χειραγωγήσουν μια σύνολο όπως η δική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυρία Φέγγ γνώρισε την αναγκαστική άβλωση. Αυτή η απάνθρωπη πρακτική θα πρέπει να καταδικαστεί όπως και όλες οι πρακτικές που εμποδίζουν τις γυναίκες να αποφασίσουν ελεύθερα κατά πόσον θα αποκτήσουν ή όχι τέκνο. Τα διαδίκτυο ε, ασχολήθηκε με το, ζήτημα και, με το ζήτημα και έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην ε, Κίνα. Η Κίνα είναι ένα κράτος 1,3 ε, δις εκατομμυρίων ψυχών. Οι αρχές της Κίνας ε, είναι έτοιμες ε, να αναθεωρήσουν τη θέση τους. Ας τους ενθαρρύνουμε να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βέρζια. Κυρία Βερζιά, δέχεστε μια μπλε κάρτα τον κύριο Είστε πολύ ευγενικοί που αναφέρατε ότι η γυναίκα έχει κάθε δικαίωμα να διαθέτει το σώμα της κατά το δοκούν. Όλοι είμαστε ιδιοκτήτες των μελών μας. Θεωρείτε λοιπόν ότι το έμβριο είναι, είναι άνθρωπος Ευχαριστώ πολύ κύριε Βερζιά. Αγαπητέ συναδελφοί, η συζήτηση αυτή για το έμβριο είναι ένα παλιό ζήτημα. Είμαι υπέρ των γυναικών να διαθέτουν ελεύθερα το κορμί τους, διατηρώ την άποψή μου και εσείς να έχετε μια αξιοπρεπή στάση σε θέματα ε, επίγοντα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορείτε να τα χειραγωγείτε και να τα εκμεταλλεύεστε για λόγους πολιτικούς και πολιτικάντικους. Ε, πρόκειται για γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους στην Κίνα λόγω ε, νομοθεσίας που δεν εφαρμόζεται. Να τις σεβαστούμε. Μην προσπαθείτε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση, τη σημερινή, να εισαγάγετε μια άλλη συζήτηση που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Vielen Dank, Frau Kollegin Herr hat Ευχαριστώ. Έχει συμπληρωματική ερώτηση ο κύριος Πόσελτ. Κυρία Βερζιάτη, δέχεστε. Παρακαλώ, κύριε Πόσελτ. Φίλε. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Δεν σας καταλαβαίνω καθόλου. Δεν ε, ε, διαστρεβλώνουμε τίποτα. Θέλω να ρωτήσω κάτι και να επαναλαμβάνω. Πιστεύετε ότι ένα αγέννητο παιδί στον 7ο μήνα, επαναλαμβάνω, στον 7ο μήνα, σε όλη την, ένεση, ε, Ένωση υπάρχει συνένεση. Στον 7ο μήνα δεν έχει δικαίωμα στη ζωή να γεννηθεί. Δηλαδή, για φανταστείτε, ένα γέννητο παιδί 7 εγκυμοσύνης δεν έχει δικαίωμα να έρθει στη ζωή. Δεν θανατώσαν τη μητέρα, το έμβριο θανάτωσαν, τη έκαναν ένωση, ε, συγγνώμη, ένεση, δηλητήριο. Είστε σαφέστατος, συνάδελφε θέλετε δικαίωμα στη ζωή του εμβρίου και είστε ε, πολέμιος της άβλωσης. Εγώ είμαι υπέρ του η γυναίκα να διαθέτει το κορμί της κάτω δοκούν. Η γυναίκα αποφασίζει και δεν πρόκειται οι άντρες να τους επιβάλλουν τι θα πράξουν με το κορμί τους. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Ε, μέχρι εδώ ήταν οι συντάκτες και τώρα ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Εσάια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική του ενός παιδιού που ασκεί η Κίνα έδειξε το της πρόσωπο για μια ακόμη φορά με την αναγκαστική άμβλωση μιας 7 ε, μηνών εγγύου. Δεν μπορούσε να πληρώσει το πρόστιμο, ήταν ήδη στο νοσοκομείο, γι' αυτό ε, έγινε όλη αυτή η ιστορία. Παραβιάζει η Κίνα τα άνθρωπα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών. Η πολιτική του ενός παιδιού αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, μόνο ε, στην επαρχία μπορεί να ε, αποκτήσει δεύτερο παιδί μια γυναίκα και όχι στις πόλεις. Εκατομμύρια όμως παιδιά, επειδή τα κορίτσια ήταν έμβρια δηλαδή θύλα, ε, θανατώθηκαν με τον τρόπο αυτό, με την άμπλωση, την αναγκαστική. 40 εκατομμύρια γυναίκες λιγότερες λοιπόν δεν γεννήθηκαν αυτά τα κορίτσια στη, στην Κίνα θεμελιώδεις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα από αυτά είναι να γεννηθεί ένα, ένας άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό δεν γίνεται σεβαστό. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Σένισιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κοινωνική πολιτική του ενός παιδιού ουσιαστικά είναι μια έκφραση παραβίασης ε, των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χαρακτηρίζεται από στήρωτητα, από στήρωση, αναγκαστική, αναγκαστική άμβλωση. 20% των ε, νεαρών και δεν γνωρίζουν κάτι εστί αντισύλληψη. Γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες αμβλώσεις ημερησίως. Η σεξουαλική αγωγή και τα φάρμακα, τα συλληπτικά ίσως είναι ο μόνος τρόπος τελικά για να πάψει η απάνθρωπη ομοία αυτή ε, μεταχείριση των γυναικών. Καμία κρατική αρχή δεν έχει το δικαίωμα να τερματίζει μια εγκυμοσύνη ή και να ε, επιβάλλει αναγκαστικά να ε, συνεχιστεί η εγκυμοσύνη μιας γυναίκας. Πρόκειται για, πολιταρχικό, για πολιταρχικά φαινόμενα, για παραβίαση της ελευθερίας. Οι γυναίκες ε, με τις πρακτικές αυτές ε, είτε χάνουν την υγεία τους, είτε μέχρι και τη ζωή τους, ή μπορεί να ε, αποφυθούν σε ακροτηριασμό, κακοποιούνται, σκοτώνονται. Αυξάνεται ο πληθυσμό στην Κίνα. Όχι γιατί γεννιούνται περισσότερα παιδιά εκεί, αλλά γιατί ζει περισσότερο κόσμος και οι κινέζικες αρχές πρέπει να αναστρέψουν ε, τις πολιτικές αυτές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ογιούλαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απαγωγή της Φέγγ Τσαν και στη συνέχεια η ε, αναγκαστική άμβλωση ήταν κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Εκτός από την έρευνα που έγινε από την τοπική ε, Δίκηση της πόλης, οι κινέζικες αρχές θα πρέπει να κοιτάξουν τι γίνεται και σε μεγάλο βαθμό με τέτοιες αμβλώσεις και στηρώσεις. Η, πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα ε, οδήγησε και σε παράνομες αμβλώσεις ε, με βάση την επιλογή του φίλου του παιδιού. Ακολούθησε δημόσια κατακραυγή και ε, αποκαλύφθηκε η περίπτωση τη Φρέγκ Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε αναθεώρηση και εξυγχρονισμό της πολιτικής ενός παιδιού. Ο οικογενειακό προγραμματισμό θα πρέπει να βασίζεται στον κόσμο παντού ε, στην επιλογή τη οικογένεια. Να υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση στην Κίνα για τη χρήση των αντισυλληπτικών και τη σεξουαλική διαπαραγώγηση των νέων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούλαντ. Κύριε Σλούτερ, μπορούμε να σα βοηθήσουμε, αγαπητέ συνάδελφε. Yes, but look that you do not lose your luggage. Ναι, αλλά προσέξτε, μην χάσετε και εσεί την αποσκευή σα κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ε, κάτι απίστευτο και φρικτό ε, συνδυασμό ε, ανάλγητους υπαλλήλους, άκαρτους υπαλλήλους που καλούνται να εφαρμόσουν μια απαράδεκτη νομοθεσία. Αυτή η πολιτική της Κίνας για το ένα παιδί ένα οικογένεια είναι Δία που φέρει τη σφραγίδα του κράτους. Μια κυβέρνηση, αν θέλει να ελέγξει τον πληθυσμό της, δεν μπορεί να το επιβάλλει δια της βίας σε καμία περίπτωση. Και τις αποφάσεις για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τον αριθμό των παιδιών, αυτό είναι μια υπόθεση των γονιών. Μπορεί το κράτος να βοηθάει, να διαπαιδαγωγεί, να ενημερώνει, ε, να ε, ε, παροτρύνει και υλικά ακόμα τον πληθυσμό. Αυτό το θέμα της αναγκαστικής άβλωσης ε, δημοσιοποιήθηκε χάρη στο διαδίκτυο, πρέπει να πούμε. Αλλά δεν είναι καθόλου μεμονωμένη αυτή η οικογενειακή τραγωδία στην Κίνα. Αν ισχύει ότι η ίδια η Κίνα ομολογεί ότι γίνονται τέτοιες ε, πράξεις και ε, ότι είναι ανήθικες, θα πρέπει και εμείς να το καταδικάσουμε και να ζητήσουμε να αλλάξει η κατάσταση και να απαιτήσουμε να δράσει εκείνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Όμπερμαγερ για ένα μισή λεπτό. Μικρό. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Μάλιστα. Ε, μας συγκινεί όλους αυτό. Δεν μπορεί να μας αφήνει ασυγκίνητους. Στον 7ο μήνα έγκαιος την απήγαγαν οι αρχές του τόπου και την ανάγκασαν να κάνει άμβλωση. 40.000 ε, γιουάν είναι το πρόστιμο. 5.000 ευρώ δεν μπορούσε να το πληρώσει. Την έπιασαν και μετά από τρεις μέρες πέντε άνδρες την, ε, ε, της έκαναν μια ένεση για να πεθάνει το έμβριο. Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη πράξη. Και δεν είναι μεμονωμένο αυτό. Από το 1979 ε, με την πολιτική του ενός παιδιού ε, ε, δεν έχουν γεννηθεί 400 εκατομμύρια παιδιά με πρόστιμα χρηματικά και με καταναγκαστικά μέτρα τις οδηγούν σε αμβλώσεις. Τι θα γίνει, εμείς θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν είμαστε σοβαροί θα πρέπει να ε, μποϊκοτάρουμε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα μέχρι να σταματήσει το Πεκίνο αυτή την απάνθρωπη πρακτική και την πολιτική του ενός παιδιού. Να την άλλαξε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ομπεμάγια. Μέχρι εδώ ήταν οι ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες, τώρα είμαι μονομένη. Κύριο Σόνικ. Το ζήτημα των ε, αυλώσεων είναι όντω ε, ένα φρικτό γεγονό. Πρέπει να καταπολεμηθεί πάση θυσία. Έμβρια δολοφονούνται. Αυτό είναι απάνθρωπο και απαράδεκτο. Μία έγκυος γυναίκα αναγκάστηκε να υποβληθεί σε άμβλωση η αυστηρή πολιτική ενός τέκνου επιβάλλεται με δρακόντια μέτρα. Και αυτό ε, τίποτα δεν μας εγγυάται πως δεν θα επανελειφθεί στο μέλλον, θα συνεχιστεί παρόμοια πρακτική. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πολιτική ενός τέκνου είναι κάτι το οποίο ε, απορρίπτεται από, τον πληθυσμό αλλά οι, οι γυναίκες πραγματικά πολλές φορές στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής χάνουν και τη ζωή τους με τις αναγκαστικές ε, αμβλώσεις. Ευχαριστώ κυρία Αντζελίλη. Ε, Πρόεδρε, στην Κίνα η πολιτική του ενός τέκνου οδήγησε σε έλεγχο των γεννήσεων μέσω καταναγκαστικών μέτρων ε, μεταξύ αυτών και την αναγκαστική άμβλωση. Όποιος, ε, όποια γυναίκα συλλαμβάνει τέκνο εκτός των ποσοστώσεων ε, δεν σε επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα και τιμωρείται με φυλάκιση καταλή, μπορεί να φτάσουν ακόμα και στην καταστροφή ε, της κατοικίας τους. Είναι απάνθρωπο να, να αναγκάζουμε μια γυναίκα σε διακοπή κοίησης μόνο και μόνο επειδή δεν έχει μια διοικητική άδεια ο πλευρά της κυβέρνησης. Θα ήταν λοιπόν περιφρονητικό να το ε, περιγράψουμε ως απλό τραύμα στην Κίνα και αυτό δεν είναι τυχαίο σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας οι γυναίκες καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών σε σχέση με τους άνδρες. Μια κοίηση που διακόπτεται θα πρέπει να ε, κληθεί ως ε, παιδοκτονία. Ευχαριστώ. Κυρία Αντζελίλη, η κυρία Σκριτλεύσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που θα εγκρίνει σήμερα θα εκφράσει την άποψή του για ε, την πολιτική της Κίνας ε, για τις αμβλώσεις. Η πολιτική του ενός τέχνου είναι ε, σαφέστατη κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση και της ακεραιότητας του, της ακαιρεότητας του σώματος της γυναίκας. Δεν μπορούν να ασκούνται τέτοιε πιέσει και να εκφοβίζονται οι γυναίκε και να ξαναγκάζονται σε άμβλωση. Είναι απάνθρωπη πίεση αυτή σε μελλοντικέ μητέρε. Γνωρίζουμε τις περιπτώσεις και μάλιστα στην Ευρώπη το 70 με 80% των ευρείων σε τόσο προχωρημένη κοίηση ε, θα μπορούσαν να γεννηθούν και να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σκριτλεύσκα. Ερχόμαστε στη διακασία ΚΑΤΣΙΑΗ και εδώ έχουν ζητήσει το λόγο πολύ περισσότεροι από όσοι δικαιούνται και από όσοι έχουν προβλεφθεί. Και θα περιστώ και πάλι στους συναδελφούς που δεν έχουν πάρει ακόμα το λόγο. Λοιπόν, ο συνάδελφος Γκάλερ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν η πολιτική του ενός τέχνου οδηγεί σε καταναλωτικέ αμπλώσει, αυτό είναι καταδικαστέο. Ε, είτε υπάρχει άνωθεν εντολή, είτε απλώς νομίζουν οι δράστες ότι του καλύπτει το κράτος. Το διαδίκτυο ε, θα φροντίσει κάτι τέτοιο να μην συγκαλύπτεται πλέον. Επίσης θετικό είναι ε, ότι θέλουν να ε, πληρώσουν αποζημίωση οι αρχές και να τιμωρηθούν οι, ε, οι θύνοντες. Ο κόσμος στην Κίνα όμως δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε τα παγκόσμια οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε να ζητήσει προστασία από το κράτος είναι μεγάλος ο κατάλογος. Ε, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, Falun στα Lao Gai, τους στέλνουν στα αναμορφωτήρια, στρατόπεδα αναμόρφωσης στη Βετιανή και πολλοί άλλοι. Καλό είναι που το συζητούμε και που επιζητούμε και διάλογο με την Κίνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλε. Η κυρία Σαμπόρσκα. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ο κόσμος έχει συγκλονιστεί μαθαίνοντας τι κάνουν οι Κινέζοι. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή η περίπτωση που μας απασχολεί. Και το θέμα αυτό είναι σημαντικό να το θέσουμε υπόψη των Κινέζων στις διμερείς μας ε, συνομιλίες. Ποιο είναι ο πραγματικό λόγο τη απαγωγή και τη αναγκαστική άμβλωση τη γυναίκα αυτή, Είναι η πολιτική οικογενειακού πραγματισμού στην Κίνα. Είναι μια κακή πολιτική που υποστηρίζεται από κονδύλια των δικών μας φορολογουμένων. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί εκείνες τις οργανώσεις ε, που υπό το πέπλο της αναπαραγωγικής υγείας προάγουν τις αμβλώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαμπόρσκα. Ο κύριος Σκίνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική του ενός παιδιού ε, της Κίνας είναι στο επικεντρό του όλου προβλήματος και το ότι επιβάλλεται μέσω αναγκαστικών αμβλώσεων. Αυτό δείχνει ε, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η πρακτική αυτή από τις κινέζικες αρχές. Είναι δική μας ε, ευχή και ξέρω ότι ε, η όλη πολιτική των ασπιθών πρέπει να εγκαταλειφθεί. Βέβαια η αναγνώριση αυτή αυτής της ε, ε, φρικτής ιστορίας επειδή δηλαδή η γυναίκα αυτή δεν πλήρωσε ένα πρόστιμο την ε, ξανάκασαν σε μετά των 7 μηνών είναι έγκυος είναι κάτι που δείχνει τελικά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση είναι στο εμπορικό παιχνίδι μέσα η Κίνα. Απλά πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν ότι πρέπει να σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζιπ. Έχει φύγει ο κύριος Τζιπ. Ο κύριος Πόσελ, τελευταίος στο Κατσιάι. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική του ενός τέκνου στην Κίνα έχει σχέση με ένα φαινόμενο το οποίο ο Σολτσενίτσιν χαρακτήρισε δικτατορία του ψεύδους, ο μέγας αυτός συγγραφέας του 20ου αιώνα. Ισχυρίζεται η κινέζικη κυβέρνηση ότι πρόκειται για μια δράση τοπικών αρχών. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Είναι συστηματική κατάσταση, γενικότερη ατμόσφαιρα εδώ και δεκαετίες. Και οι ρίζες είναι σε αυτή την πολιτική του ενός παιδιού. Και όσο ισχύει αυτή η πολιτική θα έχουμε αναγκαστικές αμβλώσεις, αναγκαστικές στηρώσεις και τέτοιες ε, βιαιότητες. Θα πρέπει να αποφασίζουν οι γονείς. Και οι γονείς, κυρία Βερζιά, είναι ο, ο πατέρας και η μητέρα, ο άνδρας και η γυναίκα. Και υπάρχει και το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού. Και αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Είναι και αυτό οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στη ζωή από τη σύλληψη μέχρι το φυσικό θάνατο. Και εμείς Ευρωπαίοι ε, να βλέπουμε λίγο τι γίνεται στη δική μας αυλή. Και ε, εδώ που εμείς δεν έχουμε εξαναγκασμούς να φροντίσουμε να μην θανατώνονται οι αγέννητοι άνθρωποι στην κοιλιά της μάνας τους. Αυτό να μην είναι παραβίαση, να μην είναι κατάχρηση ε, και για την Κίνα λέμε όχι στην πολιτική του ενός παιδιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόσελτ. <coughs> Κυρία Λούνατσεκ. Nein, nicht ναι. ναι, επί της ουσίας. Όχι, επί της ουσίας, επί της διαδικασίας. Είπατε ότι θα δώσετε το λόγο μόνο σε εκείνους που δεν μίλησαν στη σημερινή συζήτηση. Η συνάδελφος κ. Νίλσεν ζήτησε να μιλήσει στο Catch the Eye, δεν της δώσετε το λόγο, δώσατε όμως τον κύριο Πόσελτ που ήδη μίλησε. Εντάξει, μεγαλάζια κάρτα, αλλά μίλησε. Και θα παρακαλούσα να δώσετε το λόγο και στην κυρία κύριε Νίλσεν. Ευχαριστώ. Meine Κυρία Λούνατσακ, η διαδικασία Catch the Eye είναι για να γίνει συζήτηση λίγο πιο ζωντανή. Να πάρουν το λόγο και εκείνοι που δεν έχουν οριστεί από τις πολιτικές ομάδες. Η διαδικασία της γαλάζιας κάρτας είναι άλλο στοιχείο ζωντάνιας στη συζήτηση στην πρώτη συζήτηση δεν έδωσα το λόγο στο ή στον κύριο Πότσελ λόγω της κάρτας. Εντάξει, έβγαλε δύο φορές τη γαλάζια κάρτα, αποφάσισα να του δώσω το λόγο στο Κατζιά. Δεν είχε εγγραφεί από την ομάδα της. Από την ομάδα του η κυρία Κιρνίτσαν δεν είχε εγγραφεί. Τώρα χάνουμε χρόνο αντί να κερδίζουμε. Προσπαθώ να ακολουθώ μια γραμμή και πιστεύω ότι δεν κάνω διακρίσεις εις βάρος κανενός. Η κυρία Πίτροπος για να κλείσουμε. Αξιότιμα μέλη συζητάμε το ζήτημα των ε, σκανδάλου των ε, αναγκαστικών ε, αμβλώσεων στην Κίνα, στην Κίνα συμπεριλαμβανομένων και της υπόθεσης της κυρίας Φέγγ στην οποία αναφερθήκατε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησύχησε από την περίπτωση της Παντζουγιάνγκ από το Φουντσέν και από την κυρία Καρούι από το Χουλέν, που 8 και 5 μήνες έγκυες χρειάστηκε να προβούν σε αναγκαστική άμβλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε πως οι κινητικές αρχές καταδίκασαν αυτή την πρακτική και ε, εξήγηλαν ότι ξεκίνησε έρευνα και οι παραβάτες θα τιμωρηθούν. Επίσης θα γίνει μια έρευνα βρίας κλίμακος σε 19 ε, επαρχίες όπου έχουν αναφερθεί παρόμοια γεγονότα. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ε, με ε, αναφορές που αφορούν τις απειλές που αντιμετωπίζει η κυρία Φάγκ λόγω της δημοσιότητας που έδωσε στην υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες αυτές τις υποθέσεις. Τώρα, ε, αναγκαστικές αμβλώσεις και, άλλες, ε, και άλλη βία ή αλαβάναψα μέτρα κατά των γυναικών ε, που χρησιμοποιούνται στην Κίνα είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει επίσης και κάποιες παραβάσεις σε φορά τον οικογενειακό προγραμματισμό. Το συζητήσαμε το ζήτημα τον Μάιο, στι 23 Μάιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση που είχαμε στι Βρυξέλλε με τι κοινωνικέ αρχέ. Ζήτησαμε από τι Κινέζικε αρχέ να λάβουν μέτρα έτσι ώστε η εφαρμογή της πολιτικής του οικογενειακού προγραμματισμού να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον συμβάση των δικαιωμάτων. Επίσης, μας ανησυχεί το ότι ακτιβιστές, ε, πρόσωπα και, δημοσιο... και δικηγόροι οι οποίοι ε, ε, ανέφεραν αυτές τις πρακτικές και τις καταδίκασαν αντιμετωπίζουν τώρα κάποιες κατηγορίες Μετά από μια φυλάκιση της ετών ο κύριος Τσάνεν είχε τεθεί σε κατοίκον ε, περιορισμό. Το ίδιο συνέβη και με ακτιβιστές οι οποίοι αγωνίζονται κατά των αναγκαστικών αυλώσεων. Ζητάμε από τις κοινωνικές αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν ε, οι να υπερθεί η βία από πλευράς ε, των αστυνομικών αρχών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε, κύριε Χέντεγκάρτ. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος ε, ε, και ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και αρχή η ψηφοφορία. Αρχίζουμε.